Eh, Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, ισπανικά. Αν θέλετε, μπορείτε, βάλτε τα ακουστικά σας. Έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση διερμηνής που βρίσκονται σε απεργία. Βρισκόμαστε στην 24η μέρα κινητοποίησεων διαμαρτυρίας Κατά συνέπεια δεν θα παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου και η συνεδρία θα τελειώσει στη μία το μεσημέρι ακριβώ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, σύμφωνοι. Αρχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Αξιότιμα μέλη του πάνελ, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σας και να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για την προθυμία τους να έρθουν να ε, κάνουμε αυτή την κοινή ακρόαση με την Ειδική Επιτροπή ΤΑΞ 3. που συνδυάζεται η αποστολή της με τη δική μας και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση. Πριν δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές μας, ε, εμπειρογνώμονες, θα δώσω το λόγο στην κυρία Εστέρ Ντελάνγκε που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Tax 3. Οπότε θέλετε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και όπω είπατε ευχαριστώ πολύ ε, για την κοινή ε, διοργάνωση αυτή της ακρόασης συνδέοντας ε, την φορολογική απάτη και τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Είναι λίγο ασυνήθιστη αυτή η σύνδεση, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Στα τέλη του 2016 ε, διάφοροι δημοσιογράφοι της ερευνητικής δημοσιογραφίας και από τη χώρα μου, της κάτω χώρας, έκαναν ένα ρεπορτάζ που έδειξε ότι, ε, κατέδειξε ότι η Αλκάιντα ε, με ευρωπαϊκές εταιρείες είχε στήσει ένα σύστημα φορολογικής απάτης με το ΦΥΠΙΑ και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Και μετά από μεγάλες έρευνες οι ύποπτοι ε, ε, κατηγορήθηκαν ότι είχαν ε, κλέψει πάνω από ένα δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη διαδικασία ΦΠΑ. Θέλω λοιπόν να ακούσω τους εμπειρογνώμονες για να μας μιλήσουν για αυτή την υπόθεση και θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαλενθένο για να το συστήσει. Ωραία. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Μπο Έλκερ, σίγουρα κάνω λάθος στην προφορά, θα με διορθώσετε. Είστε δημοσιογράφος ερευνητικής δημοσιογραφίας, εργάζεστε ε, στην ε, κρατική τηλεόραση στη Δανία και είστε αρμόδιος για θέματα χρηματοδότησης τρομοκρατίας και ιδιαίτερα το σύστημα παρακολούθησης Echelon. Έχετε ήδη συμμετάσχει σε δημόσια κρόαση στο κοινοβούλιο μας για το Echelon οι πηγές χρηματοδότησης τρομοκρατίας συχνά είναι νόμιμες και άλλε φορές παράνομες. Κάντε λίγη ησυχία σα παρακαλώ. Οι πρόσφατε επιθέσεις κατέδειξαν ότι ε, μπορούν να σκοτώσουν με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και χωρίς κανένα κόστος πολλές φορές. Μια μελέτη που έγινε το 2015 από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Έρευνας σε θέματα άμυνας, Norwegian Defense Research Establishment, και αφορούσε την περίοδο 1994-2013, έδειξε ότι οι περισσότερες επιθέσεις χρηματοδοτούνται με λιγότερα από 10.000 δολάρια. Και ένας στους τέσσερις πυρήνες είχε χρηματοδοτηθεί από την οργάνωση που στη συνέχεια αναλαμβάνει την ευθύνη. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράση για να ενισχύσει την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τη χρηματοδότησή τη. Και ο επίτροπο Μοσκοβισή τόνισε ότι η φορολογική απάτη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το φόρο προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Θα μα εξηγήσετε σήμερα τα αποτελέσματα τη έρευνά σα, ελπίζω, ως ε, μέλος ε, της αντίστοιχης ομάδας ε, δημοσιογράφων στη Δανία και έκθεση δείχνει πως το οργανωμένο έγκλημα και οι τρομοκρατικές οργανώσεις εποφελούνται από τα ε, παραθυράκια και τα ελλείμματα που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά. Επίσης έχετε τεκμηριώσει πως οι Ισπανοί τζιχαντιστές έφτασαν στη Δανία ως επιχειρηματίες που προχωρούν με το ΦΠΑ. Θα ακούσουμε ε, την παρέμβασή σας και μετά τους συναδέλφους. Έχετε 10 λεπτά και σας ευχαριστώ που ήρθατε στην ακρόαση. Παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το όνομά μου είναι Μπο Έλκερ. Δεν είναι εύκολο το προφέρει κανεί. Είναι δανέζικο και τα δανέζικα είναι φρεχτή γλώσσα, αλλά εγώ θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Οπότε. Εδώ Θέλω να σας μιλήσω για την χρηματοδότηση μέσω της απάτης ε, ΦΠΑ και μια συγκεκριμένη υπόθεση που με την κρατική τηλεόραση της Δανίας μπορέσαμε να αποκαλύψουμε σε συνεργασία με Δανέζικη εφημερίδα και ένα σουηδέζικο πρόγραμμα εκπομπή. Ε, η υπόθεση αυτή ξεκίνησε στις 30 Μαΐου 2013 όταν συνελήφθησαν κάποια άτομα στη Μελίγια στην Ισπανία με διαφορετικές κατηγορίες ε, μεταξύ των οποίων ότι κάποιοι τσιχαντιστές είχαν λάβει μέρος σε αγώνες και δραστηριότητες στο Σαχέλ και αλλού. Αλλά ανακαλύψαμε ότι κάποιοι από τους υπόπτους διεύθυναν τρεις εταιρείες στη Δανία Και κάποιο άλλο επίση που τα απευθύνθηκαν κατηγορίε, αλλά διέφυγε, ε, είχε τη διεύθυνση μια τέταρτη εταιρεία στην Κοπενχάγη. Και οι τέσσερι αυτέ εταιρείε ασχολούνταν με αναψυκτικά και τρόφιμα και την εμπορία του. Οι συμφωνίε χρησιμοποιούνταν στη Δανία για την ε, απάτη του ΦΠΑ. Ένας άντρας επίσης καταδιωκόμενος σκοτώθηκε στο Μαλί, τον σκότωσαν ειδικέ δυνάμει γιατί ήταν υπεύθυνο μια ομάδα μάχη τη Αλκάιντα σε αυτή την περιοχή. Στην ε, περιοχή λοιπόν ε, αυτή είδαμε όλα αυτά τα άτομα που ήταν μπλεγμένα σε αυτή την εταιρεία αναψυκτικών και είδαμε πώς μπορούσαν να στήσουν αυτή την εταιρεία. Αυτοί οι Ισπανοί πολίτες μπορούσαν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δανία και με την έρευνά μας βρήκαμε και άλλους οκτώ Ισπανούς πολίτες που είχαν διασυνδέσεις με αυτήν την ομάδα στη Μελίγια και επίσης φαίνονταν να έχουν σχέση με εταιρείε στη Δανία. Όλες αυτές οι εταιρείε εμπλέκονταν σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο απάτη ΦΠΑ, σε συνεργασία και με άλλε εταιρείε, αλλά είχαν και τρομοκρατικέ προεκτάσει στην δραστηριότητά του. Είχαμε 11 άτομα ε, Ισπανού πολίτε και 24 εταιρείε, μέρο ενό ευρύτερου τρομοκρατικού δικτύου, με συστηματικέ εγκληματικέ δραστηριότητε. Το ισπανικό κομμάτι του δικτύου, βάσει τη ερευνά μα και σε συνεργασία με τη, Δανέζικα, ε, με τη Δανέζικη κυβέρνηση με 80 εκατομμύρια κορώνες, ε, σε 80 εκατομμύρια κορώνες εκτιμήσαμε ότι έφτασε η απάτη ε, που μπορούσαν να διαπράξουν σε συνεργασία εταιρείε αυτέ. Αποκαλύφθηκε αργότερα ότι τρει από τι εταιρείε συμμετείχαν και σε άλλο δίκτυο απάτη, όπου ο βασικό υπεύθυνο δικάστηκε και καταδικάστηκε στη Δανία. με 85 εκατομμύρια ε, κορώνες, δανέσκες κορώνες ποσό απάτη. Και πάλι υπήρχε ένα παρόμοιο δίκτυο στη Σουηδία που στήριζε αυτές τις δραστηριότητες. Με διάφορες κλοπέ και απάτες στο επίπεδο του ΦΠΑ. μπορέσαμε ερευνώντα ε, το πώς γίνονται αυτή οι απάτη να δούμε ότι είχε σχέση με γλυκά και αναψυκτικά, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, ε, κινητά τηλέφωνα, τυρί και κοτό κρέας πουλερικών από τις κάτω χώρες, κινητά από τη Γερμανία. Ήταν πολύ απλή απάτη του ΦΠΑ και μάλιστα κυκλικού τύπου, τύπου γαϊτανάκι τα εμπορεύματα έρχονταν από τις κάτω χώρες, μια εταιρεία που μετά διαλύθηκε και τα εμπορεύονταν με σωστά τιμολόγια, αλλά με συμπερίληψη της τιμής του ΦΠΑ που αρχικά είχε πληρωθεί και ως ε, τιμή πώλησης του προϊόντος στην πηγή. Άρα τελικά τα πουλούσαν με χαμηλότερη τιμή. Η κυκλική απάτη ήταν κάπως πιο περίπλοκη αλλά είδαμε κινήσεις του συγκεκριμένου δικτύου σε όλη αυτή την αλυσίδα. Αυτό που ανακαλύψαμε όταν είδαμε πώς αυτοί οι Ισπανοί πολίτες κινούνταν στις δανέζικες εταιρείε, είδαμε ήταν, ότι ήταν μέρος μιας ε, συμμορίας, μιας κλίκας ενός ε, τζαμιού στην Ισπανία και είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί από δύο δανούς πολίτες που είχαν ταξιδέψει στη Μελίγια ο ένα είναι Δανό πολίτη που έχασε τη ζωή του στη Συρία το 2013 και άλλο συνελήφθη αργότερα. Και οι άνθρωποι αυτοί οργάνωσαν εκεί αυτήν την ε, κλίκα αυτόν τον πυρήνα και αργότερα με την βοήθεια δαν, άλλων δανών ε, πολιτών είχαν σκοπό να εντοπίζουν δανούς πολίτες που πηγαίνουν στην ε, Συρία για να ε, δραστηριοποιηθούν εκεί. Βρήκαμε 20 Δανούς πολίτες στη Συρία και άλλοι 16 είχαν σχέση με αυτές τις εταιρείες και με το συγκεκριμένο δίκτυο. Ένας από όλους αυτούς, ένας Δανός πολίτης, ήταν ε, διευθύνων τριών-τεσσάρων εταιριών και έχασε τη ζωή του στη Συρία από, μια αεροσκάφου, από επίθεση μη επαντρωμένου αεροσκάφου το 2015. Ε, στόχος ήταν τότε ένα όχημα που ήταν επιβάτης μαζί με έναν άλλον δανοπολίτη και προγραμμάτιζαν μαζί την επίθεση στο Παρίσι. Είχαμε λοιπόν δανόπολίτη, διευθυντή εταιρεία στην ε, Δανία, που ήταν σε ένα αυτοκίνητο και προγραμμάτιζε τρομοκρατικέ επιθέσει στο Παρίσι μαζί με άλλον έναν. Ε, ο μόνος δανός πολίτης που βρίσκεται στην, στον ειδικό κατάλογο τρομοκρατίας των ΗΠΑ, τη Watch List, με ειδική παραγγελία του Σεπτεμβρίου 2013, ε, έχασε τη ζωή του από φυσικά αίτια στη Δανία. Από το 2014 μάλλον. Ε, είχε σχέσει με εταιρείε που έκανε εισαγωγέ τυριού και κινητών από τη Γερμανία και πουλερικών από τις κάτω χώρε και ε, τα πουλούσε 200 μέτρα από την κατοικία του με τρόπο νομοφανή. Στην έρευνά μας διαπιστώσαμε αλλά δεν ξέρουμε σε τι αριθμό φτάνουν, ότι υπάρχουν και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες από άλλες χώρες που μπλέκονταν σε όλη αυτή την ιστορία ένα ήταν διευθυντή εταιρεία στη Δανία και ταξίδευε από εδώ και από εκεί. Ε, τον συνέλαβαν στον δρόμο του προ τη Συρία. Η εκδίκαση τη υπόθεση του εκκρεμεί, νομίζω. Δεν είναι λοιπόν αυτό ένα πρόβλημα μεταξύ Σουηδία, Δανία και Ισπανία μόνο. Είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται με ένα δίκτυο Ισλαμιστών που αγγίζει ε, πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι δάνειοι που μπλέκονται σε αυτό το δίκτυο έχουν ε, υψηλή μόρφωση, πολλές δραστηριότητε και έχουν μπλέξει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν προεκτάσεις εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στη Δανία και αλλού. Εγώ ερευνώ την απάτη ΦΠΑ από το 2009. Μου τελειώνει ο χρόνος μου. Ναι. Α. Δεν το περίμενα. Α, δύο λεπτά. Πολύ γρήγορα τότε για να έχουμε χρόνο και ερωτήσει. Ερευνώ τι υποθέσει του ΦΠΑ από την περίπτωση του σκανδάλου του Άντροκα το 2009 όταν το μητρό άνθρακα τους Δανία χρησιμοποιήθηκε για, την, για απάτη ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας στις ανταλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Είδαμε τότε ότι υπήρχαν κάποιες χιλιάδες λογαριασμοί ε, σε ένα δίκτυο ε, απάτης ε, που χρειάστηκε να κλείσουμε τους λογαριασμούς για να καθαρίσει το δίκτυο. Όταν ερευνήσαμε ποιοι ήταν οι κάτοχοι των λογαριασμών, ήταν κάποιοι δανείοι πολίτε που έχουν σχέση με την υπόθεση του 2014 στην Ιταλία, όταν υπήρχαν υποψίε για τρομοκρατικέ προεκτάσει εκεί. Και μέσα από αυτό το δίκτυο προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Όταν εξετάσαμε τις ταυτότητές τους, είδαμε ότι έχουν πάλι σχέση με εμπορία τροφίμων στη Δανία. Πέρασαν λοιπόν από τις πιστώσεις του άνθρακα στα ηλεκτρονικά και σε άλλα ε, εμπορεύματα και στα τρόφιμα. Δεν τους νοιάζει και πάρα πολύ τι εμπορική δραστηριότητα θα χρησιμοποιήσουν ε, για να κάνουν μια πάτη νομότυπη, αλλά αρκεί να μπορεί να απολυθεί γρήγορα. Η υπόθεση στην Ιταλία συνδέεται άμεσα με την υπόθεση στην Κοπενχάγη και το ισπανικό δίκτυο. Τελείωσαν τα δύο λεπτά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να μην σας κόβουμε το λόγο. Γιατί αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά και οι άλλοι έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Ε, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρεμβολή σας. Η κυρία τώρα Ελένα Χακ η οποία είναι δικαστής και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την πρόληψη των απατών. Είστε δικαστής στην Ρουμανία, έχετε ευρεία εκπρόσωποι, έχετε μεγάλη πείρα και ήσασταν εκπρόσωπος και στην ε, ομάδα της Ευρώπης, του Συμβουλίου της Ευρώπης που δημιουργήθηκε το 1997 για την καταπολέμηση της απάτης. Έχετε μεγάλη πείρα στην καταπολέμηση των απατών και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Και είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία σας τώρα που ακριβώς κάνουμε ε, προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος. Οπότε, κυρία Χάχ, ε, σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Λέγουμε Ελένα Χαχ. Είμαι εισαγγελέα από το 1998. Έχω εργαστεί και στην Ιταλία και ήμουν και μέλος του Ανώτατο Συμβούλιο ε, Εισαγγελέων. Από το 2013 είμαι εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Και είμαι και στο Συμβούλιο του Οργανισμού στη Ρουμανία που ασχολείται με τη συλλογή προφορών για οικονομικά θέματα. Θέλουμε ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της ε, ρουμανικής αυτής αρχής και διαφόρων πηγών πληροφοριών διότι αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματο και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν τα πιστοτικά όργανα στα οποία η εταιρεία ABC έχει ένα τον Νοέμβριο του 2015 ζητήθηκαν να υπάρξει ένα έμβασμα από ένα λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό και επίσης σε ένα άλλο λογαριασμό. Οι δύο, τα δύο αυτά εμφάσματα ε, αιτιολογήθηκαν ως ε, δραστηριότητα της εταιρείας και τα ποσά ήταν από μία ζωή 150.000 από το νομικό πρόσωπο DF από ένα λογαριασμό που είχε ανοίξει σε ένα πιστοτικό ίδρυμα στη Λιβύη και υπόθηκε πως ήταν πληρωμή για εξαγωγές. Μετά από αυτό, η εταιρεία ABC δεν είχε καμία δοσοληψία πάνω των 15.000 ε, ευρώ και στους λογαριασμούς της ABC ε, βρήκαμε ύποπτα στοιχεία. Ένα μέρος των δοσοληψιών γινόταν μέσω ε, περιοχών ε, που έλεγχε το ISIS. Μεταξύ 13 και 15 η εταιρεία αυτή δεν έχει καμία δοσοληψία μέσω πιστοτικών ιδρυμάτων παρά το ότι ήταν εν λειτουργία. Η εταιρεία αυτή από το 15 έχει διάφορες ε, δοσοληψίες παρά το γεγονός ότι ένας από τους ε, ε ένα από τα άτομα θεωρήθηκε ανεπιθύμητο ένα, ανεπιθύμητο, ένα από τα άτομα που ε, ήταν αρμόδια για την εταιρεία. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η εταιρεία παρουσίασε διάφορα έγγραφα που είχε ετοιμάσει το φυσικό πρόσωπο ΤΑΒ και το άτομο αυτό ε, ε, έδωσε πληρεξούσια στον ε, πολίτη ΖΕΝΤ συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να ιδρύει εταιρείε με βάση την ομοθεσία Το άτομο αυτό ζήτα έδωσε, πληροφο... έδωσε πληροξούσιο και σε άλλο άτομο Οπότε, με βάση τα έγγραφα αυτά, οι μέτοχοι είναι το άτομο ΤΑΦ που είναι Ιρακινός και το άτομο X που είναι Λιβανέζος. Τα άτομα αυτά όμως ε, είχαν ε, θεωρηθεί ανεπιθύμητα για 15 χρόνια γιατί προπαγάνδιζαν και ε, συνέλεγαν πόρους για τζιχαντιστές. Οι δύο αυτοί αλλοδαποί βοήθησαν την παράνομη είσοδο στη χώρα ατόμων ε, που είχαν θέματα τρομοκρατίας. Αυτοί είχαν ε, ε, υποστηρίξει την παρουσία στη Ρουμανία ατόμων που ήταν ριζοσπαστικοποιημένα. Επίσης, είχαμε και άλλες πληροφορίες ότι είχαν τέτοιες δραστηριότητες. Μεταξύ 2012 και 2013 η εταιρεία ABC συνέλεξε 2 εκατομμύρια δολάρια από τη Λιβύη, τη Βουλγαρία και τα νησιά Μάρσαλ. Αυτά ε, μετατρέπηκαν σε λέει και αποσύρθηκαν ε, με, ε, ε, μέσω ταμιακών μηχανημάτων σε μετρητά. Επίσης το 2013 η εταιρεία DRP όπου είχε σχέση το άτομο T μέχρι το 2013 και οι μέτοχοι είναι ο α, και ο ζ είχαν ζωή ένα εκατομμύριο από ένα φυσικό άτομο στην ε, Συρία με την αιτιολογία ότι ήταν προκαταβολή για εξαγωγές. Αυτό μετατράπηκε σε λέει σε διάφορες φάσεις και κατόπιν αποσύρθηκε σε μέτρητα. Η συμπεριφορά των εταιρεών αυτών, ABC και DRP, είναι ασυνεπής. Οπότε μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ξέπλυμα ε, χρήματος γιατί έχουμε ε, αποσύρσεις σε μετρητά. Οπότε βλέπουμε ότι με ασυνεπή έγγραφα προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Επιπλέον υπήρχαν μια σειρά από διαδοχικά εμβάσματα μεταξύ των λογαριασμών αυτών των δύο εταιριών την ίδια μέρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή ε, αλλεπάλληλες μέρες με ακριβώς το ίδιο ποσό. Αυτά τα εμβάσματα πήγανε σε λογαριασμούς ατόμων που ελέγχουν τις εταιρείε. και η αιτιολόγηση ήταν ε, επιστροφή δανείων. Τα συμβόλαια παρουσιάστηκαν όμως ε, χωρίς ε, χρονολογική σειρά και ορισμένα ήταν ε, από το 2002 ενώ οι συναλλαγές αυτές έγιναν το 2015. Κάτι άλλο για την οικονομική δραστηριότητα έχει να κάνει με την ε, διάφορα εμβάσματα ιδίων ποσών που είναι ακριβώς κάτω από το όριο που πρέπει να αναφέρεται. Χωρίς πραγματικό οικονομικό λόγο. Αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι υπάρχει προφανής ε, πρόθεση να αυξήσει ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και να μειωθεί η φορολογία. Τα στοιχεία που έχουμε και για τη φορολόγηση και για την οικονομική δραστηριότητα για τις εταιρείε αυτές που ελέγχει ο ΤΑΦ απεκάλυψαν ότι τα χρέη προς τους μετόχους είναι λιγότερα από τους λογαριασμούς ε, συγγνώμη, από τις μεταφορές που έγιναν στους λογαριασμούς ατόμων και η συμπεριφορά αυτή θεωρούμε ότι ε, αποδεικνύει ότι υπάρχει ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματο και που έχει προκύψει από φοροδιαφυγή. Για παράδειγμα, έχουμε πολλαπλούς λογαριασμούς, μετά μεταφορές από τους διάφορου αυτού λογαριασμούς και κατόπιν ε, αποσύρσεις μετρητών και που στηρίζονται σε συμφωνίες για δάνεια ή άλλες παρόμοιες. Επίσης, τα στοιχεία που έχουμε αποδεικνύουν ότι αυτές οι εταιρείε ακόμη ελέγχονται από το άτομο T ε, μέσω ε, παρεμβολής ε, του ατόμου Z. Και ο στόχος των διαφόρων δοσοληψιών είναι να κρυφτεί ο πραγματικός δικαιούχος και να δημιουργηθεί η εντύπωση νομιμότητας. Τώρα με βάση τα χαρακτηριστικά του ατόμου ΤΑΦ και ότι έχει στηρίξει τζιχαντιστές στη Μέση Ανατολή θεωρούμε ότι υπάρχουν, υπάρχουν στοιχεία για το αδίκημα της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας μέσω της οικονομικής δραστηριότητας αυτών των εταιριών. Επίσης έχουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά το αδίκημα της ε, χρηματοδότησης τρομοκρατίας από το άτομο Z, το οποίο στη Ρουμανία ε, δρά προς όφελος του ατόμου ΤΑΦ που έχει ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητο άτομο στη Ρουμανία και μερικές σκέψεις. για να καταπολεμήσουμε ορθά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος πρέπει να συνεργαστούν πολλοί. Για παράδειγμα, τα πιστοτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί πληροφοριών, οι ερευνητές, ε, η αστυνομία και οι εισαγγελίες τα βήματα ε, πρέπει να είναι η διερεύνηση και η δίωξη. Πώς θα πρέπει να γίνεται η δίωξη της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς χρήματα. Και για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμήσουμε και τη χρηματοδότησή της. Η διευκρίνηση των χρηματικών ροών μπορεί να μας βοηθήσουν να δούμε τη δομή των ε, επιχειρήσεων αυτών να βρου, το να βρούμε πώς γίνεται το ξέπλυμα του χρήματος θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τρομοκρατία. Πρέπει να κάνουμε σωστή επιλογή, να μην πνιγούμε στα πολλά στοιχεία για, την, ε, για το ξέπλυμα χρήματος. Είναι αναγκαίο να εκπαιδευθούν ε, οι ε, ερευνητές για ξέπλυμα χρήματος, για το πώς γίνεται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Ούτε μπορούμε να διαχωρίσουμε την πρόληψη από τη δίωξη. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χακ. Είναι πάντα πολύ λίγος ο χρόνος για τόσο σημαντικές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πέντρο Σέισος Φελίσιο, τμήματάρχης στο Τμήμα Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος και Εγκλήματος κατά της περιουσίας στην Europol. Δεν είστε μόνο αστυνομικό, είστε και νομικός κύριε Φελίσιο. Εργάζεστε στη Europol, εκεί ως τμήματάρχης με ειδικότητα στα ε, οικονομικά εγκλήματα, την πλαστογραφία και τη διαφθορά. Η συμμετοχή σας ε, εδώ στην ακρόαση θα φωτίσει πολύ ένα θέμα που είναι πολύ περίπλοκο για μας ε, τώρα να λύσουμε. Θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά το πολύ και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ ενώπιον μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με χαρά βρίσκομαι εδώ και προσωπώ τη Europol. Στην εισαγωγή μου θα ήθελα να σας δώσω λίγο το πλαίσιο και να επικεντρωθώ σε τρία πράγματα. Τι κάνουμε για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τι γνωρίζουμε και ε, για τη φορολογική απάτη του ΦΠΑ και τι ποσοστό ε, είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας. Είπαμε ότι είναι κρίσιμο για όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις το θέμα της χρηματοδότησης και το χρειάζονται για να επιβιώνουν. Χρειάζονται πολλά ποσά και μόνιμη πρόσβαση σε αυτά. Το 90% όλων των τρομοκρατικών ε, οργανώσεων δεν επιβιώνουν μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας γιατί δεν έχουν χρηματοδότηση μόνιμη και ε, μεγάλη. Οι μελέτες επίσης δείχνουν ότι η Αλκάιντα στο Ιράκ ας πούμε δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν πάνω από 4 με 6 εβδομάδες χωρίς νέα φρέσκια χρηματοδότηση. Δεν έχουν καταθέσεις, δεν έχουν αποθεματικό, χρειάζονται μονίμως χρήματα ρευστά που τα χρησιμοποιούν για να καταβάλουν μισθούς. Ε, το δεύτερο που γνωρίζουμε για τις νομοκρατικές επιθέσεις είναι ότι τα περισσότερα χρήματα που χρειάζονται, τα χρειάζονται για να διατηρήσουν τις ομάδες αυτές ε, σε συνθήκες λειτουργίας. Δηλαδή, ε, η μεγαλύτερη δαπάνη είναι η μισθή. Μετά είναι η επιμελητεία, τα ταξίδια, η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η προπαγάνδα, η στρατολόγηση και κοινωνικές πρόνοιε που έχουν. Δηλαδή για τα λειτουργικά του έξοδα χρειάζονται πολύ μεγάλα ποσά. Αυτά τα γνωρίζουμε. Αυτά που δεν γνωρίζουμε είναι, για παράδειγμα, πόσα χρήματα κερδίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή για τη χρηματοδότησή του οι τρομοκρατικέ οργανώσει. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά βάσει των μελετών και των επιχειρήσεων που υποστηρίζουμε, πρέπει, μπορούμε να πούμε ότι έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση. Τη δεκαετία 85 με 95 18 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, 95 με 2005 έφτασαν στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το 2005 έως το 2016 δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες, αλλά έχουμε μια εκτίμηση για τον προϋπολογισμό για τις βασικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Και εκεί έχουν αυξηθεί τα ποσά. για την Αλκάιτα που μειώνεται τώρα και είναι στον αδύρ της 20 με 50 ε, εκατομμύρια δολάρια και για το ISIS τα περισσότερα είναι από δωρεές. Το 2015 διαφήμιζαν ότι είχαν 2 δισεκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών ε, από ε, πόρους που έχουν όταν κατέχουν κάποια εδάφη που κλέβουν τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών ή πολλούν πετρέλαιο έχει μειωθεί σημαντικά γιατί έχουν χάσει εδάφη πλέον ο προπολογισμό τους και μάλιστα έχει μειωθεί μέχρι και 80%. Αυτά τα νούμερα τι δείχνουν, ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στη χρηματοδότηση και στη δυνατότητα άντληση κονδυλίων. Από την άλλη, ε, στη φορολογική απάτη με το ΦΠΑ, τι γνωρίζουμε γι' αυτό. Είναι το μεγαλύτερο είδος απάτης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αξία. Είναι αδιανόητα τα ποσά για το μέσο πολίτη, ακόμα και για μας που εργαζόμαστε ε, στο οικονομικό έγκλημα και ε, στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είναι δύσκολο να έχουμε την τάξη μεγέθους. Και αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρούνται από τους φορολογουμένους πολίτες, αλλά ότι πηγαίνουν απευθεία σε τρομοκρατικές οργανώσεις και εγκληματικές. Είναι χρήματα που χάνει η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η παιδεία, η υγεία, βασικές υπηρεσίες και που πηγαίνει σε οργανωμένα τρομοκρατικά σχήματα και μορφώματα για να πολλούν ε, και να αγοράζουν ναρκωτικά, καπνό, διάφορες παράνομες δραστηριότητες ή ε, επενδύουν στην νόμιμη οικονομία που και αυτό είναι κακό γιατί τη διαστρεβλώνει. Και τελικά δεν επιβιώνουν οι εταιρείε που παράγουν τα καλύτερα προϊόντα ε, στις καλύτερες τιμέ, αλλά εκείνες που ε, χρηματοδοτούνται από ε, το οργανωμένο έγκλημα. Η τελευταία μελέτη έγινε το 2016 και μας λέει ότι η διαφορά του ΦΠΑ, δηλαδή το ΦΠΑ που, που συλλέγουμε σε ένα χρόνο και αυτό που θα έπρεπε να συλλέγουμε ήταν 160 δισεκατομμύρια ευρώ εκείνο το έτος και μόνο ο προϋπολογισμός της Ένωσης ήταν 155 δις. Δηλαδή, ε, εάν αποδιδόταν ο ΦΠΑ που οφείλεται, θα ήταν ένας ολόκληρος προϋπολογισμός. Βέβαια, δεν είναι μόνο η φορολογική απάτη με το ΦΠΑ και το καρουσέλ αυτό το, το καϊτανάκι, είναι 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι τεράστιο ποσό. Πόσα από τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μακάρι να ξέρα. Δεν έχουμε όμως ε, τέτοια στοιχεία, ούτε αξιόπιστες μελέτες για να το τεκμηριώσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι βεβαίως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η φορολογική απατηρία στο ΦΠΑ είναι πολύ περίπλοκα, ε, ε, δύσκολα στην κατανόησή τους και γίνονται με μεγάλη μυστικότητα και εχεμήθεια. Η απάτη ε, ε, με το ΦΠΑ ε, αποδίδει δισεκατομμύρια, χρειάζονται δισεκατομμύρια οι τρομοκράτες για να λειτουργήσουν. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Για ποιο λόγο το πιστεύουμε αυτό. Βασιζόμαστε στο έργο των συναδέλφων που διερευνούν και τα δύο αυτά θέματα, τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας και την απάτη στο ΦΠΑ. Γνωρίζουμε από πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια ποιε είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δηλαδή οι παράνομες, γιατί οι νόμιμες δεν είναι δική μας υπόθεση, με, κατά σειρά σπουδαιότητα, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, απαγωγές για λίτρα, εκβίαση ή επαναστατικό φόρος, ανάλογα πώ θα το πείτε, διάφορες δραστηριότητε λαθρεμπορίου και ε, κάθε είδους απάτη, ε, κλοπές και μικροεγκλήματα μικρή παραβατικότητα. Αυτό είναι στη δεύτερη κατηγορία χρηματοδότησης και συνολικά με όλε τι άλλε απάτες που κάνουν κατά των τραπεζών, ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικών εταιριών κτλ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα του ΦΠΑ, αλλά δεν είναι το πρώτο. Επίσης, για ποιο λόγο. Γιατί μα το λένε οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτές τις φορολογικέ απάτες με το ΦΠΑ. Αυτές οι ομάδες έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν μια δράση 10 ετών και πλέον. Οι εταιρείε αυτέ ε, είναι κατά εξακολούθηση, α πούμε, παραβάτε. Και γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί, ποιε είναι αυτέ οι ομάδε. Είναι συνήθω Γάλλο-Ισραηλινοί και Βρετανο-Πακιστανοί η έδρα τους ε, και η ηγεσία τους ε, λειτουργεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Ε, αλλάζουν και εμπορεύματα βεβαίως τα οποία χρησιμοποιούν για τη φορολογική απάτη Αλλάζουν και εταιρείε, τραπεζικούς λογαριασμούς. Καμιά φορά χρησιμοποιούν και το ίδιο δίκτυο και βέβαια όταν ε, κάποιος ε, θεωρούν ότι τον υποπτεύονται, αλλάζουν και τους ε, εμπόρους. 80% όλων των κερδών συλλέγουν και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ας πούμε, στα τρόφιμα, στη χαλιβουργία, στα ηλεκτρονικά, στα κινητά, ε, ε, στα αυτοκίνητα και τώρα έχουν ανακαλύψει και την ενέργεια. Και έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ πιο εύκολο γιατί δεν χρειάζεται να στέλνουν πουθενά προϊόντα. Λοιπόν, τα προϊόντα ήταν πολύ δύσκολο γιατί κυκλοφορούσαν προϊόντα. Οι υπηρεσίε όμω δεν χρειάζεται να στέλνονται στι παραγγελίε. Ε, στέλνουν τιμολόγια μόνο και παρέχουν την υπηρεσία. Και φέτο ήταν η μεγαλύτερη απάτη αυτού του είδους με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουν ε, ανακαλύψει και το ίντερνετ και τις επικοινωνίες voice-over και επενδύουν εκεί. Είναι επαγγελματίες χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν ε, αυτοί οι εγκληματίες. μπορεί να συνδέονται με κάποιους συλλαμιστές, εξτρεμιστές, αλλά είναι χαμηλή αυτή η ε, πιθανότητα. Έχουμε μια ιεραρχία, ε, την ηγεσία που έχει και την, πρώτη χρηματοδότηση και που διευθύνει. Μετά έχουμε τους διαχειριστές, ας πούμε, τους μάνατζερ που συντονίζουν όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε το μεσαίο επίπεδο ε, που τους ε, έχουν ως βιτρίνα ε, στις εταιρείε και το κατώτερο επίπεδο που υπογράφουν, είναι αχυρά άνθρωποι, υπογράφουν τα έγγραφα. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας γίνεται στο χαμηλότερο επίπεδο και στο μεσαίο. Δηλαδή, εκείνοι που υπογράφουν τα έγγραφα και πληρώνονται φάπαξ. Ε, Γιατί οι περισσότεροι ξένοι μαχητέ παίρνουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να πάνε να πολεμήσουν. Και αυτοί που είναι στο μεσαίο επίπεδο, ε, που είναι υποτίθεται οι έμποροι, και παίρνουν ένα μικρό ποσοστό που περνάει από την εταιρεία. Όχι όλη την απάτη. Ε, τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν στους μάνατζερ και στους ηγέτες. Δηλαδή, 2 με 10% περίπου ε, είναι ε, αυτά που παίρνουν οι διευθυντές των εταιριών. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που γνωρίζουμε και από τις δομές που έχουμε καταλήξει ότι ένα μικρό κλάσμα μόνο ε, της απάτης του ΦΠΑ πηγαίνει στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Άρα δεν θα πρέπει αυτό να μας ανησυχεί γιατί είναι πολύ μικρό το κλάσμα. Ε, όχι βέβαια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανησυχούμε, γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα εδώ, για τους δύο εξή απλούς λόγους. Ο πρώτος αναφέρθηκε ήδη από εσά. Ότι είναι πολύ φτηνές οι επιθέσεις, δηλαδή αρκεί να χρησιμοποιήσουν μόνο 10% των κερδών για να κάνουν τις επιθέσεις. 75% όλων των επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχαν ένα κόστος κάτω των 10.000 ευρώ. 600 ευρώ περίπου ήταν η απόπειρα στο τρένο Θαλής. Ας πούμε, στην Ίκαια ε, το φορτηγό ας πούμε, που έπεσε πάνω στον κόσμο είχε πολύ χαμηλό κόστος. Ε, χρησιμοποιούν ε, όπλα από την πρώην Ιουκοσλαβία. Ένα καλάσνικο 847 κάνει 400 ευρώ, μια χειροβομβίδα 50 και ένα περίστροφο 150. Ε, ακόμα λοιπόν και ένα χαμηλό ποσοστό του 60, των 60 δις είναι πολλά λεφτά, δηλαδή μισό της 100 ε, είναι 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι σεβαστά τα ποσά και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο από την 11η Σεπτεμβρίου στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά από να γίνει. Γιατί είναι δισεκατομμύρια τα ευρώ που χάνονται από την ευρωπαϊκή οικονομία ενώ αρκούν μερικές χιλιάδες ευρώ για να γίνει μια επίθεση μεγάλης κλίμακας. Συμπέρασμα, πρέπει να βελτιώσουμε τα συστήματα και την ανείχνευση. Αλλιώς ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Σήμερα σας ευχαριστώ που καλέσατε τη Europol και ε, ήρθαμε να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και για τη μόνιμη συνεργασία της ε, Europol με την Επιτροπή μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάριους Κρίστιαν Φρούντζα, που είναι διευθυντής της εταιρείας Schwarzwald Capital, που είναι μια εταιρεία οικονομικής, ε, οικονομικών συμβουλών και ερευνών. Ο κύριος Φρούντζα είναι εμπειρογνώμων στα διεθνή χρηματοπιστωτικά και δίνει συμβουλές σε τράπεζες για προδιαγραφέ αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων. Η πείρα του θα είναι πολύ χρήσιμα όχι μόνο για να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ, αλλά και για να καταλάβουμε με τι τρόπο ο ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα οι τράπεζε μπορούν να έχουν κίνητρο για να στηρίξουν τι ενέργειε των ρυθμιστικών αρχών. Οπότε οι συστάσει σα θα είναι πολύ χρήσιμε για την εργασία μα και φυσικά ε, χαιρόμεθα για αυτέ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη του πάνελ. Θα ήθελα να μιλήσω αγγλικά. Θα ξεκινήσω μιλώντας για τρομοκρατία, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Άρχισα να ερευνώ από μία, θα έλεγα, μακροπροπτική το τι συμβαίνει με το ΦΠΑ και το οργανωμένο έγκλημα περίπου από τα χρόνια της αγοράς του άνθρακα και των δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό που συνέβη από εκείνη την σκοπιά είναι ότι υπάρχει μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν τα τρομοκρατικά δίκτυα και η αλλαγή αυτή συνέβη μετά το 2010, μάλλον τη δεκαετία 2000-2010. Αυτό που άλλαξε είναι ότι με το Patriot του 2003 όλες οι τράπεζες και οι εταιρείε οι χρηματοοικονομικές κοιτάζουν πάρα πολύ την πηγή των ε, εσόδων, είτε είναι offshore είτε inshore και από πού προέρχονται ε, οι περιουσίες. Το να χρηματοδοτηθεί λοιπόν η τρομοκρατία γίνεται πιο περίπλοκο από ό,τι ήταν ε, πριν από 20 χρόνια. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μεγάλα σχέδια και δομέ με την εμπλοκή πολλών χωρών χρειάζονται και μεγάλα ποσά για να χρηματοδοτηθούν. Έχουμε λοιπόν μια νέα μορφή τρομοκρατία που θα την ονόμαζα Uber τρομοκρατία, υπερτρομοκρατία δηλαδή. Ε, και ε, έχει να κάνει με το χαμηλό κόστος, το ότι τα κέρδη παράγονται αλλού και χρησιμοποιούνται αλλού από εκεί που παράγονται. Δεν είναι η ίδια η ιεραρχία όπως στην Αλκάιντα ή στη Χεσμπολάχ ή στον ε, στρατό της Ιρλανδίας των Ρεπουμπλικάνων τότε, τον Ήρα. Ε, πώς γίνονται λοιπόν όλα αυτά. Αυτή η τρομοκρατία της Uber είναι ένα δίκτυο. Ένα χαλαρό δίκτυο. Κόσμος από τη Δανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν έχουν κάποιο κοινό συμφέρον ε, για εγκληματική ή μη δράση, ε, μπορούν να συνεταιριστούν, να οργανωθούν χωρίς να υπάρχει αναγκαστικά η διοργάνωση από μια υψηλότερη αρχή. Έπειτα το θέμα είναι πώς χρηματοδοτείται όλο αυτό. Η μεγάλη αλλαγή στην ε, τρομοκρατία αυτή τύπου Uber είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο πολύ πλούσιο από κάπου που να στέλνει χρήματα, μια μεγάλη οικογένεια, α πούμε, αλλά ο κόσμο βρίσκει, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν τα ποσά ε, κοντά του, εκεί που έχουν και την τρομοκρατική του δράση. Επίση, αυτοί οι χαμηλό κόστο τρομοκράτε, ακριβώ το χαμηλό κόστο ε, εντοπίζουν ε, και στι ανάλογε ενέργειε. Δηλαδή από, τα, από τις δράσεις ε, υψηλού κόστους περάσαμε στα χαμηλότερο κόστος, όπως το Μπατακλάν ε, στο Παρίσι. Και Περνάμε λοιπόν από την υψηλότερη ιεραρχία στη χαμηλότερη ιεραρχία, για τη μεγάλη προβολή στα μέσα μαζική ενημέρωση. Το θέμα είναι λοιπόν πώ διεργανώνονται αυτοί στη χώρα που δραστηριοποιούνται. Με πολλού τρόπου. Ε, με την απάτη ΦΠΑ, με, το, ε, με τα κρυπτονομίσματα, με πολλού τρόπου μέσα από την δράση του στου τραπεζικού λογαριασμού. Εάν δούμε του δείκτε αξιολόγηση, έχουμε όλε τι ε, μορφέ διοργάνωση. Έχουμε οργανώσει κλασική τρομοκρατία Ε, με τον, ε, με, την, με με το Ισλαμικό κράτος, να στρατολογεί ανθρώπους ε, από την Βρετάνη της Γαλλίας, ας πούμε. πράγματα περίεργα από τον απελευθερωτικό στρατό της Βρετάνης. Ε, οι τρομοκράτες θέλουν οργανωμένο έγκλημα και κοιτάζουν στα δίκτυα ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίου όπλων. Αυτό συνέβαινε περισσότερο στο παρελθόν. Τώρα το οργανωμένο έγκλημα κοιτάζει να απευθυνθεί στους τρομοκράτες. Οι διοκτικές ε, αρχές αναζητούν πλέον άλλες από τις κλασικές όδους που χρησιμοποιούσε το οργανωμένο έγκλημα. Οι τρομοκράτες δεν ε, συνδέονται αναγκαστικά μεταξύ τους με ιδεολογικές ε, ε, προεκτάσεις. Μπορεί στη Συρία να είχαν ξεκινήσει τις επαφές τους, επειδή έχει και ασφαλείς λιμένες με λιγότερες φορολογικές αρχές, δίωξη και ούτω καθεξής. Να στραφώ όμως και στο θέμα της ακρόασης αυτής, το ΦΠΑ πριν από δύο χρόνια εκπώνησα μια μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είδα ότι ένα από τα πράγματα που εμπόδιζαν την ε, ε, ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτό το κενό, το χάσμα στο ΦΠΑ. Εάν δεν υπήρχε, θα υπήρχε καλύτερη ε, ολοκλήρωση. Μιλάμε για 16 έως 18% του συνόλου των φορολογικών εσόδων στις 28 ε, χώρες μέλη. Αυτό είναι η απώλεια που έχουμε από το ΦΠΑ, ε, συμπεριλαμβανομένη στις Βρετανίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι λοιπόν δομικό κομμάτι των προπολογισμών των κρατών μελών και εκπροσωπεί εκατοντάδε δισευρώ. ευρώ. Το θέμα είναι γιατί συμβαίνει αυτή η απάτη. Γιατί χρησιμοποιούν τον ΦΠΑ, γιατί είναι εύκολο να ε, χρησιμοποιηθεί. Μπορεί κανεί να πάρει τα κέρδη αμέσω και σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα τρομοκρατών οι άνθρωποι αυτοί επικοινωνούν εύκολα μεταξύ του, ε, ανταλλάσσουν εύκολα ιδέε και είναι εύκολο να κάνει κάτι κανεί στη Δανία, να το επαναλάβει στην Ισπανία και να πάει κι αλλού. Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι τι θα περιμέναμε να δούμε στα αριθμητικά στοιχεία. Εάν ε, δούμε τι ε, ανακαλύψαμε στη Σουηδία, το Βέλιο και τη Δανία, τις βασικές υποθέσεις ε, απάτης ΦΠΑ, σε κλίμακα ευρωπαϊκή έχουμε περίπου 42 εκατομμύρια ευρώ Και εδώ δεν συμπεριλαμβάνουμε τα περίφημα ε, έγγραφα του Αφγανιστάν, που ήταν ένας άλλος ε, τρόπος χρηματοδότησης, με μεγάλες μεταφορές. 42 ε, εκατομμύρια λοιπόν. Με την τρομοκρατία τύπου Uber, όπως έλεγα. Μερικά στοιχεία, μερικές λεπτομέρειες. Πολλοί από αυτούς που εμπλέκονταν σε αυτές τις υποθέσεις διαφυγής ήταν Βορειοαφρικανοί, Ασιάτες ή από τη Μέση εκεί όπου το εμπόριο είναι παράδοσή τους. Το να ανοίγουν επιχειρήσεις, μαγαζιά ή καταστήματα ή να πουλάνε πράγματα είναι μέσα στην ε, κουλτούρα τους. Ήταν εύκολο λοιπόν να διαλέξουν αυτή την άγουσα. Επειδή όμως ο, η χρειάζεται να προσλάβει κάποιους, το ίδιο χρειάζεται και, το και ο ΦΠΑ, δηλαδή ε, ένας διευθυντής εταιρεία δεν μπορεί διαρκώς να κάνει τα ίδια, χρειάζεται νέο αίμα, νέο κόσμο που θα προσλαμβάνει και θα στρατολογεί. Υπάρχει επίσης ε, η φάση της εκμάθησης όταν αυτός που τα ξέρει τα μαθαίνει στους καινούριου ε, για να πάρουν το κολλάι των διάφορων πρακτικών. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε χώρες όπως το Ισλάμ με, με, Ισλαμ, με μουσουλμανική θρησκεία και εξτρεμιστικούς ε, και εξτρεμιστικές τάσεις συνήθως ο ΦΠΑ που επιβάλλει η κυβέρνηση δεν προηγείται του φόρου που πληρώνει κανείς στους θρησκευτικούς ηγέτες πρώτα πληρώνεται το θρησκευτικό φόρο και μετά τον ε, ΦΠΑ. Οπότε ε, έτσι βλέπουν τον ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές. Και μετά το θέμα είναι και οι διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει ε, ένα σημείο που συναντιούνται, διασταυρώνονται αυτοί που κάνουν απάτες ΦΠΑ με το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα ψάχνει νέα, νέες δεξόδους για να ξεφύγει από την προσοχή των διοκτικών δυνάμεων και της αστυνομίας. Αυτό ο τομέα λοιπόν του ΦΠΑ του προσφέρει έναν ασφαλή λιμένα, όπω λέμε. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι το μοντέλο όπως το αντιλαμβανόμαστε για το οργανωμένο έγκλημα και πώ χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλέ ε, ε περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες μεταξύ τους η μια από την άλλη. Αλλά πρόκειται για ένα παζλ με πολλά διαφορετικά κομμάτια που έχει πολλές διαφορετικές ε, προεκτάσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών και ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Ε, το ίδιο και οι σχετικέ υπηρεσίε τη τράπεζα, οι ιδιοκτικέ αρχέ επίση πρέπει να συνεργάζονται και οι εφοριακοί, οι υπάλληλοι τη οι υπεύθυνοι των φορολογικών αρχών. Δεν μπορεί κανεί να διερευνεί μόνο το ΦΠΑ ή μόνο το οργανωμένο έγκλημα και ξεχωριστά την τρομοκρατία. Πρέπει να υπάρξει μια διεπαγγελματική προσέγγιση. Και το τελευταίο είναι ότι η τρομοκρατία τύπου Uber είναι μια παγκόσμια απειλή, απειλή για όλου. Ε, Συνεχώ υπάρχουν εντάσει ε, μεγαλύτερε, αλλά αν δεν κάνει μια οργάνωση όπω το Ισλαμικό κράτο ε, η διεύθυνση και το management, όπω λέμε, επιτόπου γίνεται από ρωσόφωνους. Οι χαμηλόβαθμοι έρχονται από βορειοαφρικανικέ χώρες και χρηματοδότηση και επιμελητία από την Ευρώπη. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι ότι για τέτοια φαινόμενα ε, που είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα, ε, που εμπλέκονται πολλές περιοχές, ε, του κόσμου από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ομοσπονδία της Ρωσίας και άλλες υπήρους ε, πρέπει να συνεργαστούν όλοι μεταξύ τους. Αυτά. Και θα σταματήσω εδώ την παρουσίαση μου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμα για τις συστάσεις μας αυτά. Και τώρα να καλωσορίσω και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο μου τον κύριο Γέζεκ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Τάξε 3 και θα αναλάβει την Προεδρία Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα έχουμε πεντά λεπτά ερωτήσεων. Η ερώτηση θα πρέπει να κρατήσει ένα λεπτό και τέσσερα λεπτά για την απάντηση. Και αν υπάρχει χρόνος μπορεί να γίνει και συμπληρωματική ερώτηση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους συζητητές. Βλέπω εδώ τους συζητητές της τάξη 3. Ο Λούντεκ Νίτερμαϊερ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σε αυτή την κοινή ακρόαση, θαυμάσια ιδέα. Αναβερθήκατε στο κόστος και τα προβλήματα που έχουμε και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτές θα είναι ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, θα βοηθούσε. Σε τι βαθμό. Αυτά βέβαια θα συζητήσουμε στη δεύτερη ακρόαση, αλλά θεωρείτε ότι θα βοηθούσε. Η ερώτησή μου όμως κυρίως ασχολείται με τα διάφορα άλλα σημαντικά όργανα που είναι σε φάση εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα τα μητρώα για τους πραγματικούς δικαιούχους που θα έχουν, μας δίνουν καλύτερη πληροφόρηση. Και η σχεδόν ε, παγκόσμια ε, ανταλλαγή πληροφοριών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Θα βοηθήσουν αυτά. Δεύτερον, οι συναλλαγές σε μετρητά ε, στο παρελθόν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της εγκληματικής δραστηριότητας. Αλλά τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχουμε αυτούς τους Uber τρομοκράτες. Παίζουν ακόμη σημαντικό ρόλο οι συναλλαγές σε μετρητά και είναι σημαντικός παράγον κινδύνου. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε Ποιος ε, θα απαντήσει πρώτος. Ο κύριος ε, Σέισος. Ευχαριστώ. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Υπενθυμίζω ότι όταν δημιουργήθηκε το σύστημα υποτίθεται πως θα ήταν προσωρινό. Άρα νομίζω ότι έχει ήδη ε, περάσει την ημερομηνία λήξης του. Καλύτερα θα ήταν να αλλάξει το σύστημα. Και θα δούμε τώρα αν θα λειτουργήσουν καλά. Θα λειτουργήσουν πάντως καλύτερα από το παρόν σύστημα γιατί έχουμε μάθει από το παρόν σύστημα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μεταρρύθμιση. Για τα μητρώα αυτά, για τους ε, πραγματικούς δικαιούχους, πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει γιατί οι εγκληματίε που χρησιμοποιούν εταιρείε και λογαριασμούς για εγκληματική δραστηριότητα θα χρησιμοποιούν ε, τους ε, αφανείς ε, δικαιούχους και τους ανθρώπους βιτρίνα για να αποφύγουν την, ε, τον εντοπισμό τους. Πρέπει λοιπόν οι κυρώσεις να είναι αυστηρές και ότι οι τράπεζες θα κάνουν πραγματική έρευνα για να βρουν τους πραγματικούς δικαιούχους και όχι αυτούς που πάνε εκεί και υπογράφουν ένα χαρτί. Η πληροφόρηση για τους παγκόσμιους λογαριασμούς, ε, η παγκόσμια πληροφόρηση για τους λογαριασμούς, μακάρι να ήταν πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τις υπεράκτης και τους φορολογικούς παραδείσους Εκεί γίνονται οι τεράστιες αυτές απάτες. Αυτοί που έχουν τη γνώση και τα μέσα θα συνεχίσουν να αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες για να αποφεύγουν την επιτήρηση της Ένωσης και των διοκτικών αρχών. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε τέτοιου τύπου πληροφόρηση. Και όταν φτάνουμε σε αυτή την πληροφόρηση, φτάνουμε με καθυστέρηση 6-8 ε, μηνών και έχουν πάει σε άλλο φορολογικό παράδεισο τα χρήματα. Και μέχρι να φτάσουμε σε αυτόν έχει πάει αλλού. Ο χρόνος που κρατάνε οι έρευνές μας είναι πολύ μεγάλος. Βεβαίως, το χρήμα είναι βασιλιάς για το ξέπλυμα και την τρομοκρατία. Ο ευκολότερος τρόπος για να μεταφερθούν χρήματα, ανώνυμα, γρήγορα, αποτελεσματικά, είναι μετρητά, μέσω μετρητών. Βλέπουμε βαλίτσες ε, με χαρτονομίσματα να κυκλοφορούν. Κουτιά, πάμπερ. Και Ξέρουμε ότι υπάρχουν για παράδειγμα αυτές οι αποσκευές καμπίνας όπου μπορείς να βάλεις μέχρι 5 εκατομμύρια σε μετρητά. Και τα πιάνουμε καμιά φορά στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Τα κρύβουν μέσα σε υπολογιστέ επίση, τα μετρητά, σε γλυκά μέσα, σε φρούτα μέσα. Το οργανωμένο έγκλημα φυσικά τα χρησιμοποιεί, αλλά μάλλον και η χρηματοδότηση τη Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα συμπληρωματική ερώτηση. Όχι, να συμπληρώσω. Για τα μετρητά. Το ισπανικό δίκτυο με τους Δανούς που συνελήφθη στην ε, Ισπανία ως ηγέτης, συνελήφθη με 100.000 ε, μετρητά πηγαίνοντας στην Ισπανία. Φυσικά τα μετρητά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Και για τα δίκτυα δικαιούχων έψαχνα μια εταιρεία που είχε κάνει ένας δανός ε, ξένος μαχητής όλα τα έγραφα, όλα τα στοιχεία για την διοκτησία ήταν στο όνομά του αλλά μόνο ένα τσεκ για κάποιο νίκη είχε να κάνει με ένα λογαριασμό ενός ατόμου που ξέρουμε ότι είναι κεντρικό σε αυτή την απάτη. Μόνο απλώς, μόνο μία δοσοληψία για ένα μήνα νίκη μας έδωσε αυτό το στοιχείο. Άρα ένα μητρό πραγματικών δικαιούχων θα βοηθήσει, αλλά δεν θα επιτρέψει πραγματικά να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ και εσείς θέλετε να πείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι πολυτεχνική συζήτηση και θα μιλήσω ρουμάνικα. Για το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Προφανώς πρέπει να υπάρχει καλύτερη και ταχύτερη διασύνδεση μεταξύ αυτών των μητρών. Γιατί επειδή το επίπεδο του οικονομικού εγκλήματος και η επιδεξιότητά του για να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία υπερβαίνει τα σύνορα. Γι' αυτό τα αποτελέσματα των ερευνών είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσει ουσιαστικά την τέταρτη οδηγία που προβλέπει αυτό το Μητρό. Πρέπει να σα ομολογήσω ότι η Ρουμανία δεν την έχει εφαρμόσει ακόμη. Για εμά, για του ερευνητέ και του εισαγγελεί, το αναμένουμε με αδημονία αυτό το Μητρό εδώ και καιρό. Και ελπίζουμε το προσεχές φθινόπωρο να έχουμε τη δυνατότητα επιτέλους να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το Μητρό για να λαμβάνουμε τις αναγκαίες πληροφορίες. Τώρα για την ε, παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα και διαδικασίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Τα όπλα που έχουν οι δεν είναι τα ίδια από κράτος σε κράτος. Ενώ, για παράδειγμα, οι οργανισμοί ε, διερεύνηση οικονομικού εγκλήματος έχουν άλλες διαδικασίες. Θα έπρεπε να έχουμε ένα νέο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μην κάνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις σε πάρα πολλούς ε, προσκεκλημένους ομιλητές, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Ο Γεπ Κόφουτ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, είναι εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ ε, για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Δύο σύντομα. Πρώτα απ' όλα στον ε, συμπατριώτη μου, Πρόκειο, Στη γραπτή σας απάντηση είπατε ότι η διαπλοκή μεταξύ των, ε, η διασύνδεση μάλλον των φορολογικών αρχών, ε, της οικονομικής αστυνο, της αστυνομίας, η δίωξη οικονομικού εγκλήματος, τις αστυνομικές αρχές, ε, εμποδίζεται από τον κατακαιρματισμό των δραστηριοτήτων. Ε, και τη γραφειοκρατία. Μπορείτε να μα πείτε παραδείγματα γραφειοκρατία που κάνουν αποτελεσματική τη δράση του και την ίδια ερώτηση θέλω να απευθύνω και στη Europol. Ε, τα συζητάμε αυτόν τον καιρό. Ε, εάν πάω στη Europol, στην Εθνική Αστυνομία, τι επαφή μπορείτε να έχετε εσεί και επικοινωνία μεταξύ σα για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες εύκολα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι σε πολλές αυτές τις υποθέσεις βλέπουμε το διασυνοριακό στοιχείο αφορούν ε, πολλές χώρες ταυτόχρονα. Χρειάζεται λοιπόν ένα δίκτυο αποτελεσματικό αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Άλκια. Η υπόθεση που περιέγραψε είχε να κάνει με ένα ισπανικό δίκτυο. Η απάτη ΦΠΑ είχε ξεκινήσει το 2011. Ένα σημαντικό χρονικό σημείο. Η ομάδα δανών τζιχαντιστών που πήγαν στο Μαλί, στο Μαλί και ριζοσπαστικοποιήθηκαν παρακολουθούνταν από τις μυστικές υπηρεσίες της Δανίας από το 2006 κιόλας. Ταξίδεψαν στην Ισπανία το 2008. Η απάτη ξεκίνησε το 2011. Το 2014 οι Ισπανικές αρχές πήγαν στις Δανέζικες και ζήτησαν πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς. Πρώτη, πρώτα αντιληφθήκαμε την απάτη εκτό των μυστικών υπηρεσιών στη Δανία από την ε, Υπηρεσία Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματο. Ε, καταλάβατε τι είπα στα Δανέζικα. Είναι φρικτή γλώσσα τα Δανέζικα, σα το ξανάπα. Ε, από τον Ιούνιο του 2013 λοιπόν ήταν γνωστό αυτό ε, στην ε, Υπηρεσία Διεξουσίου Οικονομικού Και είχαν πληροφορίες για μια από τις βασικές εταιρείες από τον Ιανουάριο του 2014. Η Ισπανική ομάδα συνελήφθη τον Μάιο του 2014. Η Guardia Civil πήγε, η χωροφυλακή πήγε και του συνέλαβε τον Ιούνιο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015 Του είπα ότι πρέπει να στείλουν επίσημο αίτημα για πληροφορία. Τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε η Υπηρεσία Διεξούς Οικονομικού Κλίματος να συνεργάζεται με τι μυστικέ υπηρεσίε για το θέμα τη απάτης αυτή. Δεν ήξερε όμω ότι η υπηρεσία, οι μυστικέ υπηρεσίες τα ήξεραν ήδη το 2006 για αυτήν την ομάδα και το 2015, λίγο αργότερα, η ομάδα αυτή ε, καταγγέλθηκε στις αρχές από την εφορία όταν η εφορία έξερε να αντιλαμβάνετε τι συμβαίνει με την υπόθεση αυτή. Και πήγαν και στι μυστικέ υπηρεσίε για να πάρουν πληροφορίε για του ανθρώπου αυτού, αλλά δεν έλαβαν ποτέ πληροφορίε. Ένα παράδειγμα του πώ η γραφειοκρατία μπορεί να παρακολύσει μια έρευνα. Έρευνα που αν είχαν ξεκινήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίε νωρίτερα μυστικέ υπηρεσίε και αστυνομία, θα είχαν βρει πολύ νωρίτερα αυτά που έπρεπε. Η απάτη διαλευκάνθηκε το 2016, όταν αυτό το δίκτυο Ισπανικών εταιριών ε, που εξαρθρώθηκε. Και κάποιος που μετέφερε ένα μεγάλο ποσό σε ευρώ συνελήφθη κάποια στιγμή στην Ισπανία. Ε, έτσι λοιπόν μπορεί να δυσκολέψει την διερεύνηση μιας υπόθεσης η γραφειοκρατία. Ευχαριστούμε κύριε Σέισαρ. Η γραφειοκρατία, η απομόνωση των υπηρεσιών, η έλλειψη συνεργασίας. Αυτές είναι οι βασικές ε, Περιοχέ που θα πρέπει να μα αποσχολήσουν. Χρήζουν τι προσοχέ μα για να βελτιωθούν. Ε, στη δική μα υπηρεσία την ε, την FAU στην Πολ, έχουμε ε, ήδη ένα δίκτυο που απασχολεί διάφορους συνεργάτες οι οποίοι είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους και χρειαζόταν αυτό στη Europol. Βεβαίω, στο ανώτερο επίπεδο τη Europol λαμβάνονται διαφορετικέ ε, αποφάσει. Βεβαίω, ε, σε ανώτερο επίπεδο στη Europol γίνεται αυτή που ονομάζουμε διαγώνη επαλήθευση πληροφοριών. Δηλαδή, συνδυάζουμε πληροφορίε από τι εθνικέ υπηρεσίε των κρατών μελών με αυτά που έχουμε εμεί στα χέρια μα για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Βεβαίω, όλα αυτά δεν λειτουργούν ακόμη άψογα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ε, πληροφορίε 28, από 28 εφαγιού ταυτόχρονα, αλλά πρέπει να πάρουμε ίσως και πληροφορίες από τις αστυνομίες, τις εθνικές αστυνομίες των κρατών μελών. Δεν θα μας ενδιαφέραν οι εθνικές υποθέσεις, μας ενδιαφέρει αυτό που αφορά ε, περισσότερες από μια χώρες. Εκεί είναι η δυσκολία ε, στο να συνδυαστούν όλα αυτά γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσχέρειες και πολιτικές καμιά φορά. Ε, χρειάζεται λοιπόν περισσότερη διερεύνηση η δυνατότητα αυτή. Δηλαδή, όλε αυτέ οι πληροφορίε που βρίσκονται διασκορπισμένε από τη μια υπηρεσία στην άλλη, κάποια στιγμή να συγκεντρώνονται σε κεντρικό επίπεδο για να μπορούμε να τα διαλευκάνουμε. Για την αστυνομία και τι εφορίε τη φορολογική αρχέ πρέπει να συνεργάζονται. Λόγω των ε, νόμων και των κανόνων για το φορολογικό απόρριτο η αστυνομία πληροφορείται μόνο κάποιες υποψίες για τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ, αλλά πολύ καθυστερημένα. Ε, ήδη αφού το πρόβλημα μπορεί να ταλανίζει τις φορολογικές αρχές επί χρόνια προηγουμένως. Ε, Μόνο τότε λαμβάνει γνώση η Ευρωπούλα, αφού πρώτα ενημερωθεί και η Εθνική Αστυνομία. Έχουμε κάποια ε, παραδείγματα από τα κράτη-μέλη, τα οποία ονομάζουμε ομάδες ε, κόμπερ ε, εκεί που συνεργάζονται οι φορολογικές αρχές με την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά χρειάζονται ειδικέ υπηρεσίες στα κράτη-μέλη για την ε, διερεύνηση και την πρόληψη της απάτης ΦΠΑ με εφορία και αστυνομία να εμπλέκονται και εισαγγελεί και δικαστικούς. Είναι δύσκολος χώρος, είναι δύσκολος να τον χειριστεί κανεί αν δεν είναι ειδικό Κυρία Χακ, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γραφειοκρατία και την ερώτηση που κάνατε. Που δυσκολεύει και ε, διακυβεύει τη συνεργασία των ε, δικαστικών. Έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ε, κυκλοφορεί η πληροφορία πολύ γρήγορα για τα οικονομικά και αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τις έρευνες. Πολύ γρήγορα λοιπόν φτάνουν στους ενδιαφερομένους ε, εισαγγελείς αλλά και στην αστυνομία. Το δίκτυο αυτό και το κύκλωμα είναι πολύ πιο γρήγορο από της Διεθνής ε, αιτήσει δικαστικής συνδρομής, που είναι ένα βαρύ σύστημα, το επίσημο αυτό. Ε, η αίτηση δικαστικής συνδρομής και παροχής ε, αμοιβαία έθνους βοήθειας είναι πιο βαριές διαδικασίες. περιλαμβάνουν διάφορα αντικειμενικά στοιχεία που ξεπερνάνε τη βούληση του δικαστή που επιθυμεί μια πληροφορία. Υπάρχει αυτό το δίκτυο λοιπόν η FUNET που μας παρέχει πληροφορίες αλλά δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως αποδεικτικό στοιχείο. Γι' αυτό χρειάζεται επίσημη οδός με τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής κλπ. Το EFUNET λειτουργεί, αλλά δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, ως αποδεικτικά στοιχεία στην ε, ανάκριση. Γι' αυτό θα πρέπει να ασκηθεί πίεση, να χρησιμοποιήσουμε τους μοχλούς που έχουμε στη ε, διάθεσή μας και τα επίσημα κανάλια. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει. Επειδή είναι τεράστια τα ποσά, ε, περίπου όσο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ετήσιος. Ε, αυτά είναι χρήματα που παραδίδουμε στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες. Για ποιο λόγο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν ενέκριναν την πρόταση μεταρρύθμισης του ΦΠΑ που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκκρεμεί εδώ και ένα χρόνο και πλέον. Γιατί ανθίστανται κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπάρχουν κάποιοι κυβερνώντες που το αποτρέπουν αυτό. Αν τα εγκληματικά δίκτυα είναι τόσο ισχυρά και τόσο πλούσια, δεν αποκλείεται τίποτα. Πώς εξηγείται αυτή την αντίσταση των κρατών μελών να, κλείσουν αυτό το παραθυράκι που επιτρέπει να ε, λειτουργούν οι εγκληματίες. Όλο για την ασφάλεια μιλούν οι κυβερνήσεις, αλλά αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν το λύνουν. Για ε, τα μετρητά, όπως είπε ο κύριος Έσος, Φελίσιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, αλλά πώς προχωρεί αυτή, προχωρεί αυτή η υπόθεση. Υποτίθεται ότι το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ θα έπρεπε να καταργηθεί. Όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, του έκανε αυτή την ερώτηση. Ε, είναι ειδική περίπτωση, αλλά δεν είναι η μοναδική. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν. Και επίσης θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τα κρυπτονομίσματα. Εσείς μιλήσατε για αυτά κύριε Φρούνσα. Η Μάλτα και άλλες χώρες, όχι μόνο η Μάλτα. μπαίνουν στο κρυπτονόμισμα και προβάλλουν και ε, προωθούν ε, την επικράτειά τους ως μια χώρα που μπορεί κανείς να κάνει business σε κρυπτονόμισμα. Ποιος θέλει να απαντήσει. Κανείς ε, δεν τολμάει να κάνει κάποιες εικασίες. Το δεύτερο, για το θέμα των μετρητών, ο κύριος Φρούντζα. για τα κρυπτονομίσματα. Ε, όχι, αργότερα. Τώρα για τα μετρητά, δεύτερη ερώτηση. Έγινε μια ερώτηση ειδικά σε μένα. Yeah. Okay. So... Α, να το πω. Ναι. Όπως γνωρίζετε τα κρυπτονομίσματα είναι μια υποκατηγορία των ε, ψηφιακών νομισμάτων που γεννήθηκαν στη δεκαετία του 90. Ε, και εκτός από το PayPal τότε έκλεισαν όλες οι πλατφόρμες για ξέπλυμα χρήματος. Πολύ γρήγορα πέρασαν όλοι στο κρυπτονόμισμα. Όλοι ε, γι' αυτό μιλάνε, δεν ξέρουν τι είναι. Είναι πάνω από 1500 νομίσματα. 249 κράτη αλλά λιγότερα νομίσματα. Στην Ευρώπη έχουμε 4-5 νομίσματα μόνο παγκοσμίω. Αλλά ε, στο διαδίκτυο έχουμε 1500. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τόσα πολλά νομίσματα. Τι κάνει πια ο κόσμο και θέλει τόσα πολλά νομίσματα. Υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι είναι εγκληματική δραστηριότητα και δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό πλέον, είναι, έχει αποδειχθεί. Υπάρχει διαδικασία αυτή mining, δημιουργία νομισμάτων, ε, ε, που είναι πολύ κερδοφόρα. Μπορεί ο καθένας να παράξει χρήμα. Και ως φυσικό πρόσωπο δεν χρειάζεται να είσαι καταχωρισμένη εταιρεία στην Ευρώπη ε, ίσως με την εξαίρεση της ε, Μάλτας και των χωρών της Βαλτικής. Αλλά κανονικά μπορεί ο καθένας να το κάνει από τον υπολογιστή του. Και αν αναρωτηθεί κάποιος από πού προέρχονται τα νομίσματα, Εγώ μπορώ να, κόψω ας πούμε νόμισμα Μονέρο ή ε, bitcoin. για, ποιο λόγο το κάνει κανείς αυτό. Γιατί την πηγή εισοδήματο αφενός και αφετέρου μπορείς να στείλεις χρήματα παγκοσμίω παντού σχεδόν, εκτός τραπεζικού συστήματος. Και αυτό είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Το δε κόστος, να περάσεις από κρυπτονόμισμα σε υλικό νόμισμα είναι 9% περίπου, δηλαδή σε, χαρτονομίσματα. Αλλά σήμερα πολλοί ακόμα και για την παροχή, για υπηρεσιών δέχονται και ε, κρυπτονομίσματα, όχι φυσικά νομίσματα. Αυτό, να καταλάβετε τι σημαίνει για να περάσουμε και στα μετρητά ή ακόμα για τα κρυπτονομίσματα. Ναι, για τα κρυπτο μπορώ να πω κάτι. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Το 2014 ήρθα στην Europol και θα σας έλεγα ότι όλα αυτά είναι κατασκευάσματα και δεν υπάρχουν τέτοια κρυπτονομίσματα. Φυσικά τα πάντα αλλάζουν ραγδαία και οι ίδιοι τρομοκράτες και υπήρξαν περιπτώσεις ε, πλατφορμών crowdfunding ε, στο διαδίκτυο ε, που ανοιχνεύτηκε ότι συνδέονται με εξτρεμιστές, Ισλαμιστές και φυσικά συλλέγουν από εκεί χρηματοδότηση. Λίγες περιπτώσεις, τρεις-τέσσερις, δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι απάτη που χρησιμοποιήθηκαν χρήματα για λότριους σκοπούς, πάντως το διαφήμιζαν και ορισμένα τα κονδύλια που συνέλεξαν από την μαζική αυτή χρηματοδότηση είναι αυτού του τύπου. Επίσης πάλι στο διαδικτύο οι τρομοκράτες μεταξύ τους εκπαιδεύουν ένα τον άλλον με εγχειρίδια, πώς δημιουργούνται, πώς αγοράζονται, πώς πολλούνται αυτά τα νομίσματα με οδηγίες χρήσεως είναι ακόμα στην αρχή αυτή η προσπάθεια, δεν τη θεωρούμε μεγάλη απειλή, αλλά εκπαιδεύονται και αφιερώνουν χρόνο σε αυτό. Επίσης, το γνωρίζουμε επειδή είναι πολύ εύκολο να μεταβιβαστούν αυτά τα χρήματα με ένα τηλέφωνο, με ένα φορητό υπολογιστή παντού, αν έχει ε, ίντερνετ. Και ορισμένοι ξένοι μαχητέ χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για να μεταφέρουν ε, τα χρήματα από την Ευρώπη στις εμπόλεμες περιοχές όταν μεταβαίνουν εκεί. Είναι πολύ μικρό βέβαια αυτό. Ε, αλλά χρειάζεται προσοχή και μεγάλη γιατί είναι και ε, καινούριο στο οργανωμένο έγκλημα. Εδώ και χρόνια το χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι ναρκωτικών και τα λοιπά. Ας πούμε για τα καρτέλ στην Κολομβία έχει γίνει συνήθις πρακτική. Πέρυσι ε, πήγαμε και διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιούν ε, μαζικά τα κρυπτονομίσματα, τα καρτέλ, τα κολομβιανά. Για να μεταφέρουν την αξία που παράγουν από ε, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία. Και υπάρχει τεράστια αύξηση ε, από τον ένα χρόνο στο άλλο. Έχουν εξοικειωθεί, δεν τα φοβούνται πια αυτά τα συστήματα ως νέα και άγνωστα. Ε, άλλη ερώτηση για τα μετρητά. Την ίδια ερώτηση, τη δεύτερη, θέλει κανείς να την απαντήσει. Ε, είναι από τα προσφυλή μου θέματα αυτό το θέμα των μετρητών. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει πολλά από την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, βεβαίως μέχρι τα τέλη του έτους θα σταματήσουν να τυπώνουν τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, αλλά τουλάχιστον 20 χρόνια ακόμα θα κυκλοφορεί νόμιμα ε, το χαρτονόμισμα. Στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Οι εγκληματίε προσπαθούν να ξεφορτωθούν αυτά τα χαρτονομίσματα γιατί δεν το κατάλαβαν. Πηγαίνουν στις τράπεζες και ε, ε, αλλάζουν και καλά κάνουν γιατί καταφέραμε να πιάσουμε μερικούς έτσι. Κάποιοι άλλοι που το κατάλαβαν κάνουν το αντίθετο τα αγοράζουν και πληρώνουν περισσότερο από την ονομαστική τους αξία, 15% παραπάνω, γιατί ξέρουν ότι είναι καλή επένδυση, γιατί είναι εύκολα στη μεταφορά και ε, εύκολα μεταφέρονται. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Παραμένουν λοιπόν τα μετρητά στις μεταφορές. Ευχαριστώ. Από την Άλτε. Um, Καρολίν Πικό. για το κυβερνοέγκλημα, γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί την Europol μια ερώτηση. Πώς άλλαξαν οι προτεραιότητες και τα μέσα σας τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσετε το νέο τους νέους τρόπους απάτης και τα εικονικά νομίσματα και αν θεωρείτε ότι οι ενέργειες της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, για παράδειγμα η οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος και η οδηγία για το ΦΠΑ, βοηθούν, θεωρείται ότι βοηθούν κάτι γενικότερο. Η διμερή συμφωνία που έχουμε με την Νορβηγία, που νομίζω ότι εγκρίθηκε το Φεβρουάριο από το Συμβούλιο, θεωρείται ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει για να μειωθεί η απάτη του ΦΠΑ θα μπορούσε να ήταν μία μέθοδος που θα μπορούσαμε να, έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε και για άλλες τρίτες χώρες. Και αν ναι, με πιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ο εκπρόσωπος Europol. Κάναμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο από το κύβερνο έγκλημα ιδιαίτερα για τα εικονικά νομίσματα. Έχουμε το κέντρο για το κύβερνο έγκλημα, ένα αυτόνομο, με παρκές προσωπικό. με γύρω στους 140 προσωπικό. Ένα από τα κύρια καθήκοντα αυτού του κέντρου ήταν να μελετήσει και τα εικονικά νομίσματα έχουν ε, προσλάβει τους καλύτερους εμπειρογνώμονες, τους έχουμε εκπαιδεύσει εμείς, εγώ συγκεκριμένα, πηγαίνουν στα κράτη-μέλη, προσπαθούν να εξηγήσουν ε, τι γίνεται και έχουν ε, εκπονήσει και εγχειρίδια που είναι πραγματικά πρότυπα όχι μόνο για την Ένωση αλλά για όλες τις χώρες του κόσμου για τα θέματα αυτά. Είμαστε σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα, που είναι πολύ σημαντικός, βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο και για τα εικονικά νομίσματα και γενικότερα για το οικονομικό έγκλημα. Νομίζω ότι εμείς ως Europol ε, είμαστε έτοιμοι. Τώρα τα κράτη-μέλη θέλουν λίγο χρόνο ακόμη. Αλλά ξέρουμε ότι θα προκύψει, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Πολύ καλές οι αλλαγές στην οδηγία για τον ΦΠΑ, γιατί φυσικά θα πρέπει να είναι και οι ε, φορείς που κάνουν συναλλαγές με αυτά τα νομίσματα υπεύθυνοι για να δίνουν στοιχεία για την ύπαρξή τους, τη λειτουργία τους και να αναφέρουν όπως οποιοδήποτε κανονικό πιστοτικό ίδρυμα όποιες ε, συναλλαγές τους φαίνονται ύποπτες. Βεβαίως, έχουμε το blockchain, αλλά έχουμε ένα μόνο αριθμό. Πρέπει να ξέρουμε ποιο κρύβεται πίσω από τον αριθμό αυτό, άρα πρέπει να μα το δώσουν αυτοί οι φορεί. Ναι, νομίζω ότι η συμφωνία με την, με την Νορβηγία θα βοηθήσει την ενισχυμένη συνεργασία γιατί θα ανταλλάσσουμε όχι μόνο στρατηγικά στοιχεία αλλά και για προσωπικά στοιχεία θα έχουμε επαφή μαζί τους, θα τους καλούμε σε συναντήσεις. Χρειαζόμαστε τέτοιε συμφωνίες και με άλλες χώρες. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα της Europol γιατί από τότε που ε, νεκρήθη ο νέος κανονισμός. Εσείς αποφασίζετε γι' αυτά και δεν έχω τις γνώσεις που χρειάζεται για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Η κυρία Χακ. Για τα κρυπτονομίσματα. Ναι. Θέλω να κρούσω ένα διαφορετικό κόδωνα κινδύνου. Οι πλατφόρμες όπου ανταλλάσσονται τα νομίσματα αυτά είναι ίσως όνειρο για τον καθένα μας και από πλευράς κατάρτισης. Γιατί όλοι θέλουμε γρήγορο πλουτισμό. Ωστόσο, για μας τους ερευνητές αυτές οι πλατφόρμες ε, ε, μας δημιουργούν προβλήματα. Τρομερά. Είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τα άτομα που κάνουν αυτές τις συναλλαγές. Τις συναλλαγές. Ποιος αγοράει, ποιος πουλάει. Είμαι πεπισμένη. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλωσορίσουν με ενθουσιασμό την πέμπτη οδηγία που θα επιτρέπει να ελέγχονται οι συναλλαγές που γίνονται μέσω των εικονικών αυτών πλατφορμών. Στο ρουμανικό σύστημα η Κεντρική Τράπεζα επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει και τονίζει ότι δεν είναι φυσιολογικό το ότι αυτά τα κρυπτονομίσματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτή είναι μόνο η δική μας εθνική πολιτική. Αλλά δεν θέλουμε βέβαια να εμποδίσουμε το επιγραμμικό εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από το ΙΕΝΕΦ e ο Μάριο Μποργέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εισηγητές. Πρώτο σημείο. Θεωρούν μήπως οι εμπειρογνώμονές μας ότι κάτι σημαντικό ως προς την έλλειψη υποθέσεων που να έχουν διερευνηθεί για το σύστημα απάτης ΦΠΑ και γενικώς φορολογικής απάτης και φορολογικής νομιμότητας για τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας είναι κάτι που καθορίζεται από την απόλυτη έλλειψη της διαλεύκανσης τέτοιων ε, συναλλαγών και δραστηριοτήτων επειδή δεν ανακαλύπτονται από το τραπεζικό σύστημα. Ε, υπάρχει το τραπεζικό απόρριτο. Δεν έχουν πολλά σχέση με αυτό. Ξέρουμε ας πούμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα της μαφίας χρειάστηκε την παρέμβαση υψηλών ε, δικαστικών λειτουργών, υψηλών βαθμών και ίσως αυτή να είναι η αιτία που διευκολύνει την απάτη ΦΠΑ ε, σε, στη χώρα πρώτης ε, άφηξης των εμπορευμάτων όταν αυτά πηγαίνουν σε άλλη χώρα. Μήπω αυτή η τρύπα είναι το πρόβλημα και επιτρέπει αυτή την κερδοσκοπία σε σχέση με, την, με το ΦΠΑ. Επίσης για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που δόθηκαν ως παραδείγματα ε, είναι ενδιαφέρουσες και αυτή της Δανίας και για άλλες σκανδιναβικές χώρες και επειδή μερικά αφορούν υπόθεση και της Ιταλίας. Και είναι έρευνες που ξεκινούν με την ανακάλυψη μια απάτη του ΦΠΑ και τελικά καταλήγουν σε συγκεκριμένου υπόπτου, σε πρόσωπα που όπως είδαμε ας πούμε στην περίπτωση της ε, υπόθεσης της Δανίας ήταν ε, τζιχαντιστές στη Μελίγια. Δεν γίνεται όμως να γίνεται αυτό ο έλεγχος εξάντε, δηλαδή να βλέπουμε την πορεία των προσωπών αυτών που ξεκινούν από περιοχές τρομοκρατικής δράσης και μετά επιστρέφουν στην Ευρώπη και συχνάζουν σε τζαμιά. Ευχαριστώ. Ε, πρώτη ερώτηση για το τραπεζικό σύστημα. Κυρία Χάκ. Ναι, να προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για την ε, παρακολούθηση που δεν είναι απλή στα χρηματοοικονομικά δίκτυα. Ξέρουμε ότι πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου και αν υπάρχει παραμικρή υποψία χρηματοδότησης τρομοκρατίας ε, πρέπει να οδηγούν σε σήμανση όμως ακριβώς το χρηματοοικονομικό σύστημα θα πρέπει να παρακολουθείται αυστηρότατα. Μόλις ε, λάβει χώρα μια ύποπτη συναλλαγή πρέπει να σημανθει απευθεια απευθείας, όχι μετά από τρία-τρει μήνες, διότι εάν τρία χρόνια μετά ο εισαγγελέα το πάρει χαμπάρι και ε, κάνει καταγγείλει την συναλλαγή, έχει φύγει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον. Και εδώ δεν κατηγορώ κανέναν, απλώς θέλω να πω ότι αν ήταν αυστηρότερες οι κυρώσεις προς τις τράπεζες, αν ήμασταν λίγο πιο πιεστικοί, ε, και αν τελικά έχουν το περιθώριο να μην καταγγέλουν αμέσως τις υπόπτες συναλλαγές, δεν προχωρούμε. Θα έπρεπε το κάθε κάτω μέλος να λάβει Και έπειτα, αυτός που επιβάλλει ποινές και το ας πούμε ραντάρ ανακάλυψης των ύποπτων συναλλαγών θα πρέπει να είναι κάπως ανεξάρτητος και αμερόληπτος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να επιβάλλει κυρώσεις στις τράπεζες εάν αυτό αποφασίζεται από κάποιο διοικητικό συμβούλιο ας πούμε που βρίσκεται κάπου ε, σε μια κρατική υπηρεσία ή υπουργείο. Είναι προσωπική μου άποψη, είμαι βαθιά πεπισμένη, πλήρως πεπισμένη, ότι ε, ένας επόπτης, ένας ελεγκτής τραπεζών που είναι τελείως ανεξάρτητος μπορεί να αιτιολογήσει και θέλει να ε, και διαπιστώσει μάλλον ότι μια τράπεζα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια ύποπτη συναλλαγή, τότε μπορεί να επιβάλλει και ποινή. Αλλιώς δεν υπάρχουν τα σωστά κριτήρια. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να προσπαθήσει να απαντήσει. Όταν ξεκίνησα ερευνώντα την απάτη ΦΠΑ από το Δανέζικο Μητρό του Άντρακα, με τον συνάδελφό μου τότε είδαμε ότι υπάρχει ένα μητρό ανθρώπων, κατάλογος ανθρώπων που έχουν εμπλοκή σε ύποπτες συναλλαγές. Λίγοι από τους λογαριασμούς αυτούς ε, των ανθρώπων αυτών ήταν ε, τελείως νόμιμοι. Μιλάμε για περίπου 200-300 λογαριασμούς, αλλά καταλήξαμε σε 36 που μας ενδιαφέραν. Οι περισσότεροι λοιπόν είχαν σχέση με ύποπτες συναλλαγές. Όταν κοιτάξαμε αυτή την ομάδα, είδαμε μια Γαλλο-Ισραηλινή ε, ομάδα που αναφέρατε κι εσείς, ή και ομάδες ε, αγγλοπακιστανικές την Ιταλική μαφία, ε, μαφίες της Ανατολικής Ευρώπης, από το Χονγκ Κόνγκ και την Ταϊβάν ε, και άλλες συμμορίες. Πολλές τέτοιες ομάδες τύπου do it yourself. Ήταν διασυνοριακή, διαθρησκιακή και διαπολιτισμική η δράση τους. Πρόεδρος, μάλιστα. Φαίνεται ότι εκπροσωπούνται ισότιμα όλες τις περιοχές του κόσμου, λοιπόν. Και τώρα έχουμε χρόνο και για τη διαδικασία Κάτσε, Έχω τρεις ομιλητές στον καταλογό μου. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κινίτση από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας ε, και οι παρουσιάσεις τους ήταν πραγματικά διεξοδικές για το πρόβλημα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της απάτης, ΦΠΑ και τη διαπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα και τις, τις εγκληματικές οργανώσεις. Έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω και πολλές ήδη τέθηκαν, αλλά θέλω να σταθώ στο εξής. Καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένου αριθμού, αλλά πόσο επηρεάζει η παράνομη δράση των ε, ε, ομάδων εγκλήματο στην χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, διότι είναι σημαντική η σχέση των παράνομων δραστηριοτήτων, ακόμη και των κλασικότερων, ε, και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σήμερα έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να αναχαιτήσουμε και τη δράση των οργανωμένων ομάδων που όπω είπατε έχουν δράσει διασυνοριακή με στόχο πολλέ φορέ να χρηματοδοτούν τρομοκρατικέ οργανώσει. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε όμω την νομοθεσία σχετικά, διότι πρέπει να γίνει εδώ κάποιο βήμα πρόοδου. Και μετά σε ό,τι αφορά αυτά που προηγουμένω συζητήθηκαν, την FIU και την ε, διασύνδεση των εθνικών FIU για να μπορούμε να εντείνουμε τη συνεργασία τους που για την ώρα είναι κάπως κατακαιρματισμένη. Ε, και να ερευνήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θέλω να μου πούνε οι προσκεκλημένοι μας τι πιστεύουν, πώς θα σχολίαζαν την πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Απριλίου ε, κανόνες για να απλουστευθεί η ανταλλαγή πληροφοριών οικονομικού χαρακτήρα ή άλλου είδους προκειμένου να εντοπιστούν εγκληματικές δραστηριότητες χρηματοδότηση άλλων εγκληματικών δράσεων. Νομίζω ότι η οδηγία αυτή θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δίκτυα χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και κυρίω την έλλειψη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εφαγείων και των ε, αστυνομικών και διοκτικών αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την πρώτη ερώτηση παραδοσιακές μορφές ε, εγκλήματος και τρομοκρατίας. Κύριε Σέισας. Ναι. Είναι γεγονός ότι και εμείς έχουμε διαπιστώσει κάποιες αλλαγές. Ε, ιστορικά λεγόταν ότι υπάρχει ο χάσμα και διάκριση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία οι ε, ε, κλιματίες ήθελαν να κερδίσουν λεφτά στη ε, παρανομία και χωρίς προβολή, ενώ οι τρομοκράτες υποτίθεται ήθελαν να αλλάξουν πολιτικά κάποια κατάσταση με προβολή και δημοσιότητα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και στο παρελθόν η μικροεγκληματικότητα και το οργανωμένο έγκλημα συνδεόταν με την τρομοκρατία, αλλά η μεγαλύτερη σύνδεση που έχουμε διαπιστώσει είναι αυτή που συζητούμε σήμερα ο οικονομικός κόσμος και ο χρηματοπιστωτικός κόσμος. Γιατί εκεί τα πάντα συνδέονται. Το χρήμα δεν έχει ε, οσμή και η παραοικονομία συνδέει την τρομοκρατία με τον εγκληματικό κόσμο. Όταν διώκουμε το οικονομικό έγκλημα ε, βρίσκουμε και ε, τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένο έγκλημα. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ευρώπη ξεπλένουν ε, τα έσοδα από ένα ευρύτατο λαθρεμπόριο ναρκωτικών ε, σε διάφορες χώρες τα νομιμοποιούν αυτά τα, τα χρήματα και τα ξαναστέλνουν στη Λατινική Αμερική και κρατάνε ένα ποσοστό. Τα έχουμε διαπιστώσει αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλέον ε, σαφής διάκριση ε, στα οικονομικά. Είναι όλα παραοικονομία και αυτοί κυκλοφορούν ελεύθερα γιατί χρειάζονται τα χρήματα και οι δύο, και το οργανωμένο έγκλημα και οι ε, τρομοκρατικές οργανώσεις. Για την πρώτη ερώτηση θέλετε να απαντήσετε, όχι γιατί στη δεύτερη. Ωραία. Ως ε, εισαγγελέα μπορώ να πω ότι οι οικονομικές πληροφορίες που ε, παίρνουμε από τις μονάδες οικονομικών οικονομικών ε, υπηρεσιών, δίωξη οικονομικού εγκλήματο είναι πολύ σημαντικέ. Ξέρουμε ότι οι τράπεζε και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γενικώ επικαλούνται το τραπεζικό απόρριτο και είναι απρόθυμέ να δίνουν πληροφορίε στι αρμόδιε διεκτικέ αρχέ. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει τι FIU, τι ε, μονάδε ε, ε, οικονομικών πληροφοριών. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό αυτό. Και ε, ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις οικονομικές προφορίες που μας παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες και είναι για μας χαρά αυτό και μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι οι μονάδες ε, οικονομικών πληροφοριών ε, έχουν ε, διαφορετική δομή από χώρα σε χώρα. Αλλού είναι οι διοικητικέ δομές, αλλού είναι οι υβριδικές ε, δομές, αλλού εμφανίζονται ως ε, τμήμα των διοκτικών αρχών. Ε, ακόμα στη Ρουμανία παρά είναι διοικητική αυτή η δομή. Εμείς θα προτιμούσαμε υβριδικό χαρακτήρα γιατί εμείς εισαγγελεί χρειαζόμαστε ε, αυτές τις των οικονομικών αναλυτών θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ορισμένες ε, πληροφορίες όταν αναλύονται οδηγούν σε χάραξη στρατηγικής. Θέλω λοιπόν εγώ ως εισαγγελέα όλες αυτές οι μονάδες που κάνουν αυτές τις αναλύσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μοχλό και να τις κάνουν και να τα διαβεβάζουν αυτά εγκαίρως τους εισαγγελείς και τις διοκτικές αρχές. Ευχαριστώ. Uh, ε, για το σχέδιο οδηγίας για το FIU, τις ε, μονάδες ε, ε, οικονομικών πληροφοριών, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Εδραιώθηκε αυτό το δίκτυο στη Europol, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ περισσότερο, να έχουμε τους απαραίτητους πόρους να γίνεται αυτό, αλλά ποια είναι η ιδέα στη Europol. να υπάρχει μια ευρωπαϊκή δομή FIU, ε, Υπηρεσίας Οικονομικών Πληροφοριών. Ε, όχι απλώς να συλλέγουμε αυτά που μας θέλουν τα κράτη και οι αστυνομίες, αλλά να έχουμε και καλύτερα εργαλεία στη διάθεσή μας, όπως ένα σύστημα εντοπισμού της τρομοκρατίας, όπως το TFTP, τη συμφωνία που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε επίσης να έχουμε και ΣΔΙΤ με κάποιες από τις μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη για να ανταλλάσσουμε πληροφορίες ε, σε ένα περιβάλλον με περισσότερη εμπιστοσύνη. Μια αντίστοιχη προσπάθεια κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πόρους και ε, ανθρώπινους και οικονομικούς για να γίνουν όλα αυτά πιο λειτουργικά και να μπορούμε να ανταλλάσσουμε στοιχεία πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες. Συμφωνώ απολύτως. Και εμεί στο Κοινοβούλιο και στην προηγούμενη επιτροπή που είχαμε για τα έγγραφα του Παναμά, στην τελική μα έκθεση καλήσαμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις μονάδες οικονομικών πληροφοριών και ως προς του ανθρώπινους πόρους και ως προς τα χρήματα και ζητήσαμε και κάποιο είδους εναρμόνιση σε κάποιο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την τρίτη ερώτηση, για το σχέδιο οδηγία για τη χρήση οικονομικών πληροφοριών για την καταπολέμηση κάποιων εγκλημάτων. Υπάρχει κανένα σχόλιο? Όχι, πραγματικά, όχι. Ωραία. Η κυρία Γκόμες. Το να καταργήσουμε τις ανώνυμες μετοχές είναι κάτι που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας και μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο σε χώρες όπως η Ρουμανία ας πούμε. τι ξέρετε για την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση ξεπλήματος βρωμικού χρήματος και για την εγγραφή εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, υπάρχει το πρόβλημα αυτών που είναι εξωευρωπαϊκέ και έχουν επιχειρηματική δράση στην Ένωση. Αυτό το αρνήθηκε το Συμβούλιο. Αλλά πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτό τώρα να εξυπηρετήσει κάπου. Η κυρία Χακ. Ιστορικά και παραδοσιακά η μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες είναι και οι ανώνυμες μετοχές και στο σκάνδαλο του Παναμά είδαμε σχετικά δεδομένα. Ε, πολλά τέτοια στοιχεία. Υπάρχει η διεθνή στάση να απαγορευτούν οι ε, ανώνυμες μετοχές από τις περισσότερες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες γίνονται ακόμα αποδεκτές. Το είδαμε από το Panama Papers. Οπότε τι νόημα έχει να υπάρχει μια προτιμησιακή γραφή όταν κάποιοι μπορούν να πουλήσουν τις εταιρείε τους και μόνο με ένα κομμάτι χαρτί ε, και μετά δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως θα θέλει αυτό να συμβεί εδώ παντού. Βέβαια και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίω ε, στους φορολογικούς παραδείσους, ε, τα offshore όπου καταθέτουν όλα τα χρήματά τους αυτοί που θέλουν και είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο διεθνές σύστημα, αλλά θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο να καταργούνταν όντω οι ανώνυμες μετοχές. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Θα πρέπει, όπως έλεγα πάντοτε, να, είμαστε, να είναι κανείς έντιμος όταν είναι δικαστικός λειτουργός. Μπορεί τώρα να εκπροσωπώ τη Ρουμανία, αλλά είμαι Ρουμάνα δικαστικός. Και πρέπει να πω με τα θλίψεις ότι η Ρουμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι και ο καλύτερος μαθητής ε, στο σύστημα αυτό. Πρέπει να είμαι έντιμη και ειλικρινής. Η Ρουμανία δεν έχει εφαρμόσει ακόμα πλήρως την τέταρτη οδηγία. Και ως εισαγγελείς εμείς, χωρίς αυτό το μητρό των ε, δικαιούχων, των κατόχων, ε, του προτιμησιακού καταλόγου των κατόχων, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βεβαίω χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έρχεται και η πέμπτη οδηγία, αλλά καλά θα ήταν σε εμά τουλάχιστον να αρχίσει να εφαρμόζεται η τέταρτη προηγουμένω. Ω εισαγγελέας λοιπόν είμαι βεβαία ότι η πέμπτη οδηγία ε, θα προσφέρει ωφέλη. Είναι βελτίωση για τη δουλειά μα. Πρέπει όμω προηγουμένω η Ρουμανία να εφαρμόσει σωστά την τέταρτη οδηγία. Και μετά θα αντιληφθούμε και την πέμπτη. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Η Νίνα τελευταία μιλήτρια από του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν παρούσα για τις παρουσιάσεις των ομιλητών. Ψήφισα σε μια άλλη επιτροπή, ελπίζω να μην επαναλαμβάνω θέματα που ήδη καλύφθηκαν. Η κυκλική απάτη του ΦΠΑ είναι μεγάλο πρόβλημα σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε, και συγγνώμη αν επαναλαμβάνω ορισμένα που υπόθηκαν, θα ήθελα να μάθω ποιες χώρες έχουν ε, τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης και ποιες το να αντιμετώπισαν αυτή την απάτη επιτυχώς. Εστιάζουμε κυρίως στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τις τράπεζες και στις ύποπτες πληρωμές. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τομέας που δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί καθόλου. Άτομα ε, που διαμένουν σε άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσής τους εντός της Ένωσης που έχουν δικαίωμα διαμονής αλλά κάθε φορά που φεύγουν ε, εκμεταλλεύονται το σύστημα ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ε, αυτής της κατάστασης που πηγαίνουν έρχονται και υποφελούνται. Και το τρίτον, οι νέες τεχνολογίες ε, η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain μπορούν να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η απάτη ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι κυρώσεις που υφίστανται τα πιστοτικά ιδρύματα λειτουργούν αποτρεπτικά ή είναι επαρκείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις πρώτες δύο ερωτήσεις. Θα τη συζητήσουμε και στο δεύτερο γύρο συζητήσεων. Ήδη αναφερθήκαμε στα κρυπτονομίσματα ή τα εικονικά νομίσματα. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Όχι. Για τα κρυπτονομίσματα. Ο κύριος Φρούντζα. πώς να αξιοποιήσουμε το blockchain και πώς να χρησιμοποιήσουμε το blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη. Το Dubai είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία blockchain για να διευκολύνει τον έλεγχο πληρωμής του ΦΠΑ. Αν όλα ήταν ε, ε, ψηφιακά, θα ήταν λύση το blockchain, γιατί εύκολα μπορείς να δεις την ιδιοκτησία και όλη την αλυσίδα αλλά αν έχεις ένα εμπορευματοκιβώτιο γεμάτο κινητά τηλέφωνα περιπλέκεται κατάσταση. Όταν περάσουμε σε ε, απτά προϊόντα και μάλιστα σε ευαίσθητα προϊόντα, τρόφιμα κτλ. περιορίζονται δυνατότητες. Τώρα τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς ε, ήδη χρησιμοποιείται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η εφορία έχει ένα μεγάλο τμήμα για την ε, εκμάθηση των μηχανών, των μηχανών, την τεχνητή νοημοσύνη και νομίζω και σε άλλες χώρες της Ένωσης γίνονται παρόμοιες προσπάθειες. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να καταλήξει στο ότι αυτό το άτομο κάνει αυτό. Θα σου δώσει κάποιες τάσεις, μια γενική εικόνα. Στον τραπεζικό τομέα, για παράδειγμα, λένε ότι η εξόριξη δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να τα λύσουν όλα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο. Η επιτόπου εργασία επί συγκεκριμένων υποθέσεων είναι πολύ πιο απαραίτητη σήμερα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ε, ε, απάτη του ΦΠΑ, η εύκολη απάντηση είναι να καταργεί το ΦΠΑ, όπω στι ΗΠΑ. Άμα δεν έχει ΦΠΑ, δεν έχει και απάτε ΦΠΑ. Πρόεδρο, ευχαριστώ όλου του ομιλητέ μα για την παρουσία του, για τι απαντήσει του, για τι παρουσιάσει του. Πήραμε όχι μόνο μια πολύ καλή γενική εικόνα, αλλά και πολύ λεπτομεριακή πληροφόρηση, κάτι το οποίο θα επηρεάσει και τις εκθέσεις μας. Την έκθεση της Επιτροπής Τάξη 3 τουλάχιστον. Ο, η απάτη του ΦΠΑ, επειδή τα ποσά είναι δεράστια, και επειδή είναι εύκολο να διαπραχθεί, ευκολότερο από το να μπει να ληστέψεις μια τράπεζα, προφανώς ε, προσελκύει και τους τρομοκράτες και είναι σημαντική πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οπότε, έχει επιπτώσεις και στην ασφάλεια των συμπολιτών μας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην καταπολέμησή της. Όπως θα πούμε και στον επόμενο γύρο συζητήσεων που θα συνεχιστεί στα πλαίσια της Επιτροπής τάξε σε λίγα λεπτά. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Βαλενθιάνα. Απλώς να ευχαριστήσω τους ειδήμονέ μας και όλους τους συναδέλφους που είπε όπου όπως είπε ο συμπροεδρός μου μας ανέφεραν ε, πολλές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την εργασία που πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς απλώς μπορούμε να νομοθετήσουμε ουσιώδες, αλλά για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε πρέπει να ξέρουμε και τις ανάγκες και τα κενά που πρέπει να καλύψουμε. Η Επιτροπή ε, και η δική μου και η τάξη 3 μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση της νομοθεσίας και να κάνουν και πολλές άλλες συστάσεις που φυσικά θα κάνουμε και θα σας τη στείλουμε. Είναι προφανές ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πολύ ε, όλους και ιδιαίτερα τους δήμονές μας. Χαίρετε. Πρόεδρος, σε λίγα λεπτά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Τάξε 3.